ζητά τροποποίηση ε, κάποιων μελών ε, σε κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Ε, ο κατάλογος των ορισμών θα περιληφθεί στα πρακτικά και αν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι την έγκριση των πρακτικών θεωρούνται αυτές οι τροποποίησεις και ορισμοί ότι εγκρίνονται. Πέρα των ανακοινώσεων και περνάμε στην έναρξη της σημερινής συζήτησης. Παρακαλώ εκ νέου τους συναδέλφους. Έχουμε να συστήσουμε πολύ